Συνεχίζουμε λοιπόν. Είναι τιμή για μένα που προεδρεύω αυτού του τμήματος της Ολομέλειάς μας. Καλωσορίζω τον κύριο Επίτροπο. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Επίτροπο. Τα χθεσινά πρακτικά είναι διαθέσιμα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια σχόλια. Δεν υπάρχει παρατήρηση λοιπόν για τα πρακτικά. Θεωρούνται δεκτά. Το πρώτο σημείο τώρα στην ημερήσια διάταξη είναι η ετήσια έκθεση.